Dear uh, we ε, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ε, μία δοκιμή να κάνουμε, παρακαλώ. Βάλτε την κάρτα στη σχισμή. Κάντε ότι ψηφίζετε, άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ, πιέστε τα κομβία. Ναι, θα καταλαβαίνω. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. I close the vote. Τέλος. Ψηφοφορίας λειτουργεί το σύστημα. Dear friends, uh, first... Αγαπητοί φίλοι, πρώτο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι το σημείο 10 πλαίσιο για την ε, ετικετοθεσία της ε, ενέργειας ε, υπό τον κανονισμό 69F. Η συγκητής μας ο Ντάριο Ταμπουράνο ονομαστική κλίση έναρξη της ψηφοφορίας για την προσωρινή συμφωνία που επετέφθη μετά από ε, τριμερή διάλογο επί τη βάση του άρθρου 69F πέρας ψηφοφορίας. Uh, Ωραία, καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται. Το αποτέλεσμα του τριμερούς. 11. Σχέδιο έκθεσης για την ε, πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τροποποιητικός κανονισμός που αφορά την ε, προ αγωγή τη σύνδεση ε, στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες, εισηγητή ο κ. Ζωρίνιο. Ε, τροπολογία 19, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μεταφορές 16, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπολογισμός 13 υπέρ κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται 17 μεταφορές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 126 θα σας περιμένω. 126. Στο δικά μου έγγραφο είναι η σελίδα 10. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 Ρέτζι 2 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές ε, απο, ε, εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μεταφορές 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές ε, ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 57. Ελέγχουμε την 57. Έχουμε έναν παραπανίσιο από το ΕΛΚ που ψηφίζει. Εντάξει τώρα. Ωραία, ευχαριστώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 58. Και προπολογισμό 6 είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 47 υπέρ κατά αποχές ε, ε, ε, απορρίπτεται. 8 της Ρέτζη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 και 61 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τις δύο τροπολογίες από κοινού. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Τροπολογία 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ναι, έλεγχος ηλεκτρονικός. Δεύτερο τμήμα. Τέλος ψηφοφορίας. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μεταφορές 8 υπέρ κατά ας ελέγξουμε. Μεταφορές 8. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η κυρία Τόγια δεν έχει κάρτα, οπότε δεν γίνεται, ε, απορρίπτεται. Μάλιστα, οπότε έχουμε ισοπαλία. Ήταν 30 ε, υπέρ, 29 κατά. Ήταν η τροπολογία 9 τώρα. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 18... 80, 80, τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μεταφορές 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτζετ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 και μεταφορές 14 μαζί. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τρανσ, ε, μεταφορές 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελ, τελική ψηφοφορία, ονομαστική κλίση για το σχέδιο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται. Ευχαριστώ. Πέρασε τις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και ψηφοφορία για να ξεκινήσουμε τις διοργανικές διαπραγματεύσεις 69F, ε, ονομαστική κλίση, πέρας της ψηφοφορίας. Ε, γίνεται δεκτή και αυτή η εντολή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και σε όλους τους κοιόδης και σε όλη την Επιτροπή μας. Μπράβο μας. Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, σημείο 12 στον κατάλογο. Έχουμε εισηγητή τον κύριο Μπουτικόφερ. 67 και 68 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 83. Ψηφίζουμε την τροπολογία 83. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Απολογία 84 υπέρ, κατά, ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται να το ελέγξουμε. 84. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 84. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη, προσθήκη 1 στη συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Προσθήκη 1 στη συμβαστική 11. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προσθήκη 2 στη συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται μάλλον, αλλά να το ελέγξουμε. Προσθήκη 2 στη συμβαστική 11. Πέρας εφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 99. στις πληροφορίες. Απορρίπτεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 103. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 104. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 108. Πέρας. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προσθήκη 1 ε, στη συμβαστική 14 συγγνώμη υπέρ κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την προσθήκη 1 στη συμβαστική 14 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται ε, προσθήκη 2 στη συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε και αυτό ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και αυτό. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 141. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στην ε, συμβαστική 17 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την προσθήκη στη συμβαστική 17. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στη συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την προσθήκη στη συμβαστική 18. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ, 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, α, εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη 1 στη συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την προσθήκη 1 στην συμβαστική 22. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προσθήκη 2 στη συμβαστική 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Διορθώνει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται. Αλλά ας το ελέγξουμε κιόλας. Προσθήκη 2 στην συμβαστική 22. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη στην ε, συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ναι, ναι, να το ελέγξουμε. Προσθήκη στην συμβαστική 23. Πέρας πληροφορίας. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Εγώ έκανα λάθος. 2.23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ γιατί δεν βλέπω ξεκάθαρα πώς ψηφίζετε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στην 24. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Δεν είναι πολύ σαφές. Ψηφίζουμε την προσθήκη στην συμβαστική 24. Πέρας ψηφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στην 25. Υπέρ. Κατά να το ελέγξουμε ως συνήθως. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 269. Πέραση οφορίας. Απορρίπτεται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2,71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2,72. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 13 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την ΙΜΚΟ 13. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 284 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 286 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προσθήκη στη συμβαστική 31 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την προσθήκη στην συμβαστική 31. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.97 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε και αυτό. Ψηφίζουμε τη 2.97. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.27 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 327. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 325. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 325. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 329 υπέρ, κατά, αποχές να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 329. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 331 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 332 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μεταφορές 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μεταφορές 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μεταφορές 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μεταφορές 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Μεταφορές 7 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Μεταφορές 9 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Μεταφορές 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 2 υπέρ κατά να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την δεύτερη τροπολογία. Πέρας πληροφορίας, απορρίπτεται. 10 ε, υπέρ κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας πληροφορίας, Απορρίπτεται. Employment 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, απασχόληση 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 27 της Επιτροπής Μεταφορών. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Πολιτισμός 8 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 12 της Επιτροπής Πολιτισμού. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Και αυτό. Τροπολογία 13. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 6 υπέρ. Ε, κατά. Να το ελέγξουμε. Δεν είναι σαφές. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. ΥΜΚΟ 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 12 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 12 της ΙΜΚΟ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ήμικο 18 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Πέρα σου φορείας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στην συμβαστική 7 υπέρ, κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την προσθήκη στη συμβαστική 7. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μεταφορές α υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Ε εγκρίνεται. Ε, απασχόληση B. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνατε. Ένα. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Τροπολογία 1. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά. Να το ελέγξουμε και αυτό. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά. Ελέγχουμε και πάλι την τροπολογία 3. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε. Τέσσερα. Πέρα στους εφορίες. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Συγγνώμη. Αλλά δεν μπορώ να πω φως. Τροπολογία 5 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ο κύριο Έλλερ. ένα ερώτημα. Ε, ποια είναι η νομική βάση για, την, ε, για το συμβιβασμό. Ένας, μια συμβαστική πρόταση είναι το μόνο σημείο που υπάρχει νέα διατύπωση, γιατί έχουμε συμβιβασμό. Οι άλλες προτάσεις είναι ε, προσθήκες. Τι θα πει προσθήκη στο συμβεβαστική πρόταση. Είναι πολύ τυπική διαδικασία αυτή, συνηθισμένη. Συνηθισμένη είναι... Είχαμε τέτοιες προτάσεις. Όταν ψηφίζουμε μαζί με την ΙΜΚΟ, το ίδιο, οι ίδιες προτάσεις ήταν. Για την ψηφιακή ενιαγορά. Είχαμε τέτοιες προσθήκες γιατί ήταν οι προσθήκες της, ε, προστα, προτάσεις συγγνώμη της ΣΥΜΚΟ. Καταρχάς, αν μπορώ να συμπληρώσω, δεν υπάρχει ε, ούτε συντάκτης ούτε ε, ομάδα για τις προσθήκες αυτές. Και όταν ψηφίζουμε μια, προσθήκη, μια ε, συμβαστική πρόταση πρέπει να ξέρουμε το σύνολο της συμβαστικής. Όλα τα άλλα είναι συμπληρωματικές ε, ε, προτάσεις, οι οποίες όμως πρέπει να ψηφίζονται πριν την τελική συμβαστική πρόταση. Τώρα δεν μπορούμε να, κάνουμε, να έχουμε απόψη για το πώ θα είναι η τελική έκθεση. Δεν είναι σωστό να ψηφίζουμε τη συμβαστική και μετά τι προσθήκε σε αυτήν. Uh, Mr. okay. Ε, λοιπόν, συνάδελφοι, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε αυτή τη διαδικασία από κοινού με την ΙΜΚΟ, γιατί ήταν πολύ συνηθισμένη η διαδικασία για αυτούς. Όχι, έχετε δει και ότι για εμάς δεν είναι τόσο συνηθισμένη αυτή η διαδικασία, αλλά με την ΙΜΚΟ είχαμε διάφορα προβλήματα με τους και κτλ. Και, και στο τέλος αποφασίσαμε να κάνουμε κι εμείς αυτές τις προσθήκες στις συμβαστικές προτάσεις. Ναι, στο μέλλον βέβαια δεν θα κάνουμε την ίδια, δεν θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Θα έχουμε βέβαια και συνεργασία με την ΙΜΚΟ και σε άλλους φακέλους, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε αν όντως θέλει η ΙΜΚΟ να, έχει, να κάνει προσθήκες σε κάποιες α, α, προ, το, τροπολογίες. Ο κύριος Μπουτικόφερ θέλει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η διαδικασία συμφωνήθηκε από όλες τις ομάδες που παρέστησαν στις, συναντήσεις των, στις δύο συναντήσεις των σκιωδών που είχαμε οργανώσει. Η μία ομάδα που δεν παρέστη ήταν η ΕΝΕΦ. Όλες οι άλλες ομάδες συμφώνησαν με τη διαδικασία αυτή. Και η ουσία ήταν η εξής. Για κάποιες από τις συμβαστικές τροπολογίες είχαμε συμφωνία μεταξύ πέντε ή παραπάνω ομάδων. Για τις προσθήκες ωστόσο είχαμε ε, συμφωνία μεταξύ τριών ή τεσσάρων, μικρότερος αριθμός εν πάση περιπτώσει ομάδων. Και συμφωνία υπήρχε. Τώρα αν το αμφισβητήσουμε αυτό, θα πρέπει να δούμε την, ε, την, να αμφισβητήσουμε τη διαδικασία, όχι το αποτέλεσμά τη. Αν θέλετε να αμφισβητήσουμε κάτι, είχε να κάνει με τις πλειοψηφίε που δημιουργήθηκαν στην ε, συνάντηση των σκιωδών όλα το, όλο το επιπρόσθετο κείμενο που προτείνεται, προτείνεται από τουλάχιστον τρεις ομάδες οι οποίες εκπροσωπούνται στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί φίλοι, να προτείνω κάτι. Για το μέλλον. Οι συντονιστές μας θα πρέπει να συζητήσουν το θέμα αυτό πριν βεβαίω ακούσουν και τι απόψει των πολιτικών ομάδων. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε τώρα εδώ στην ανοιχτή συζήτηση, γιατί κάποιοι συνάδελφοι θα πούνε εντάξει, είναι καλή η διαδικασία, κάποιοι θα πούνε όχι, δεν είναι σωστή η διαδικασία. Οπότε καταλαβαίνω, αλλά θα το αφήσουμε για τη συνάντηση των συντονιστών. Γιατί τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη διαδικασία, επειδή ψηφίσαμε γι' αυτό. Και όπως ακούσαμε, οι εισηγητές, οι σκιώδεις, αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να το συζητήσουμε, εντάξει, να το συζητήσουμε. Η κυρία Τόγια έχει πρώτα το λόγο και μετά ο κύριος Τούρμες. Ένας-ένας, με τη σειρά. Μετά ο κύριος Κάρινς και μετά εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην πράξη η παρέμβαση του εισηγητή καθιστά άχρηστα τα λόγια μου γιατί θα έλεγα ακριβώς τα ίδια ότι αυτή η διαδικασία ήταν καρπός μιας κοινή απόφασης στην οποία, ε, όπου συμμετείχαμε ε, στις, ε, ε, και όσοι συμμετείχαν στις συνεδριάσεις των σκιωδών το γνωρίζουν και εκεί συμφωνήσαμε ότι εκεί όπου υπάρχουν σημεία ακόμα και περιφερειακά αλλά για μας σημαντικά που δεν ανέπιπταν στις συμβαστικές εμείς θα τι προτείναμε. Άρα λοιπόν θεωρώ πως όχι μόνο πρέπει να επιβεβαιώσω την εργασία του εισηγητή, αλλά και να πω ότι ήταν όλα απόλυτα σωστά και ε, χρήσιμη γιατί συμπεριλήφθηκαν όλες οι αποχρώσεις και όλες οι σύμβολες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τούρμες. Καλή είναι η πρότασή σας βρίσκω. Θα πρέπει να τη συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Όμως ναι, πρέπει να συμφωνήσω ότι συμφωνήσαμε συνενετικά για το Industry 4.0 και δεν θέλω να παρατραβήξουμε αυτό το θεσμικό θέμα. Current. Επειδή εγώ είμαι συντονιστής θα έπρεπε να είμαι ευχαριστημένο ότι θα μπορούμε να το λύσουμε σε επίπεδο συντονιστών, αλλά αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για ε, διαδικαστικό κανόνα. Και είναι θεμητό η φύση της συμβιβαστικής είναι νέο κείμενο που βασίζεται σε νέες υπάρχουσες τροπολογίες. Και εδώ το έχουμε αρκετές φορές ε, χρησιμοποιήσει εδώ και τα ψηφίζουμε σαν προσθήκες όταν είναι ε, τροπολογίες επί των ε, συμβιβαστικών. Εάν υπάρχει μια προσθήκη για μια συμβιβαστική, είτε είναι διαφορετική συμβιβαστική, είτε έχει τελείως διαφορετικό και ασαφές ε, ε, καθεστώς ε, και ποιος καταθέτει την, τροπο, την συμβιβαστική, αν ταιριάζει με τη συμβιβαστική ή όχι. Ορισμένοι θεωρούν ας πούμε ότι η συμβαστική είναι καλή αλλά χωρίς αυτή την προσθήκη και έτσι δυσκολεύει η ψηφοφορία. Τώρα εδώ είμα... χάσαμε αλλά ξέρουμε χασαμε ότι μπορούν, μπορεί να αντιστραφούν οι ρόλοι και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ε, αν θέλουμε ή όχι να χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είναι αυτό στην παράδοσή μας. Είναι θέμα όμως των συντονιστών. Πρέπει να το συζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι οι συντονιστές, οι συγητές και σκιώδεις συγητές δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τον κανονισμό επειδή ξαφνικά τους συμφέρει επειδή έρχεται ένας πράσινο συγητή, ο οποίο θέλει να περάσει κάποια πράγματα μαζί με τη συνεργασία τη αριστερά. Και αυτή η προσθήκη στον συμβιβασμό δεν είναι πλέον ο συμβασμός που ψηφίσαμε στην αρχή. Είσαστε και δυόμιση χρόνια πρόεδρο τη Επιτροπής, ε, της ε, Διάσκεψης των Πρόεδρων. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η Επιτροπή θα δεχθεί τέτοια παραβίαση του κανονισμού. Τέτοιο πράγμα δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί. Και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι και η ΙΜΚΟ από εδώ και πέρα δεν θα δεχθεί τέτοιες ανοησίες. Ούτε η ΜΚΟ, λοιπόν. Η κυρία Νίμπλερ, είναι σημαντική η σειρά, είναι σημαντική η σειρά θα λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Νίμπλερ, θα είμαι και εγώ σύντομη. Υποστηρίζω τους συναδελφούς που είπαν ότι πρώτον είναι ζήτημα κανονισμού. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να αποφασίσουν οι εισηγητές, οι ισκιώδεις, οι συντονιστές και ούτω καθεξής. Και εγώ υπήρξα εδώ, στην παρούσα Επιτροπή, πρόεδρος της Επιτροπής. Τέτοια διαδικασία δεν γνωρίζω, αλλά ούτε και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε σας ζητώ να το ξεκαθαρίσετε κάτω από τη σκοπιά του κανονισμού και να μας εξηγήσετε στο μέλλον πώς θα κινηθείτε. Να κάνετε λοιπόν εσείς την διευκρίνηση για την επόμενη φορά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ εσείς. Δεν έχει μικρόφωνο η κυρία που μιλεί. Ωραία λοιπόν. Να προσθέσω κάτι ακόμη. Εάν συνεχίσουμε την πρακτική αυτή, εδώ πρόκειται για νομοθέτημα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν ψηφίζουμε νομοθεσία, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα. Ακόμα και αν είναι έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο από πριν γιατί σε περίπτωση ψηφοφορίας για νομοθετικό κείμενο δεν μπορούμε να έχουμε την αβεβαιότητα αυτή. Δεν ξέρω τι κάνει η ΙΜΚΟ, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Ε, ξαναλέω, όταν θα πρόκειται να ψηφίσουμε νομοθετικό κείμενο. Ο Πρόεδρος. Αγαπητοί φίλοι, όπως είπα και πριν από λίγο, θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό μεταξύ των συντονιστών. Δική μου ευθύνη είναι βέβαια, το εξήγησα προηγουμένω και έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά οφείλω να σα πω ότι με του κανονισμού είναι λίγο διαφορετικοί οι κανονισμοί ανά κοινοβουλευτική επιτροπή και ούτε τα περιγράφουν όλα με απόλυτη σαφώνεια, σαφήνεια συγγνώμη, οι κανονισμοί. Για παράδειγμα το ζήτημα του bidding είναι ανάλογο με κάθε επιτροπή και αλλάξαμε και εμεί του κανονισμούς μας για την προσφορά ε, βαθμών στην, ε, πριν από ένα χρόνο περίπου. Δεν είναι απόλυτα σαφέ λοιπόν το τι λέει ο κανονισμό. Να σα δώσω παράδειγμα. Παραδείγματα μάλιστα και από τη δική μας Επιτροπή. Σας διαβεβαιώ ότι εάν δεν υπήρχε προηγούμενο στην δική μας Επιτροπή δεν θα ήμουν διατεθειμένος να δεχθώ την τρόπο του κανονισμού και να πω ότι αλλάζουμε τα πάντα τώρα στην Επιτροπή μας. Αλλά είχε συμβεί και παλιότερα. Και θα σας δώσω παραδείγματα. Θα ήθελα να τελειώσει εδώ η συζήτηση γιατί είναι απολύτως αναγκαίο να αποφασίσουμε για το μέλλον. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας. Και χρειάζονται κανόνες που να έχουν διάρκεια. Πιθανώς υπήρξαν λοιπόν οι αλλαγές αυτές λόγω Τη επιτροπή ΙΜΚΟ που αυτοί μας πίεσαν πολύ προ αυτήν την κατεύθυνση. Μπορούμε όμως εμεί να επανέλθουμε και να πούμε ποτέ πια. Μπιουτικόφερ τελευταίο. Ο κ. Μπιουτικόφερ. Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να διευκρινιστεί με κάποιο τρόπο το θέμα. Ε, εγώ δεν έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτό. Το κάναμε διότι διαμορφώθηκε συνένεση για το ζήτημα αυτό. Και κανένας από μας των, μεταξύ των σκιωδών εισηγητών δεν είχε την αίσθηση ότι παραβιάζει κανονισμούς στη συνάντηση επαναλαμβάνω των σκιωδών εισηγητών. Δεύτερο, αποκρούω την επίθεση του φίλου μου Βέρνερ Λάγκεν, ε, προσωπική επίθεση, την αποκρούω διότι λέει ότι επειδή υπήρξε ένας πράσινος εισηγητής ερχόμαστε τώρα και αλλάζουμε τον κανονισμό. Όχι, αυτό μου φαίνεται ότι είναι απολύτως άδικο Βέρνερ. Το ανακαλώ, λέει ο κ. Λάγκερ. Δεν εννοούσα άλλωστε καν τον κύριο Πιτικόφερ, άλλον εννοούσα. Ωραία, λέει ο πρόεδρο. Ε, γίνεται πολύ ιστορικό ε, στην αίθουσα. Θα λυθεί το πρόβλημα για την Επιτροπή μας. Πάντως σας βεβαιώ ότι οι κανονισμοί μας δεν είναι απολύτως σαφείς για να μπορεί κανείς να κρίνει με απόλυτη ε, ε, σαφήνεια. Ζήτησα το λόγο, ευχαριστώ που μου τον δίνετε. Πράγματι διαρωτώ με τι είδου παιχνίδι παίζουμε εδώ. Γιατί περιμένανε το τέλο τη ψηφοφορία για να φέρουν όλε αυτέ τι ενστάσει. Η συζήτηση θα γίνει στου συντονιστέ. Άρα εμεί οι ευρωβουλευτέ που ψηφίσαμε αδίκως μέχρι τώρα για το τίποτα. Αυτό σημαίνει. Α, όχι, όχι, πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Αν υπάρχει κάποια δυσκολία, αν υπάρχει κάποια διαφορά προσέγγισης τη ψηφοφορίας. Θα έπρεπε να τα είχαν πει τα πράγματα αυτά πριν να αρχίσει η ψηφοφορία. Ο πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, κλείσαμε τώρα τις ψηφοφορίες για το θέμα αυτό. Συζητήθηκε το θέμα για 15 λεπτά. Προχωρούμε στην επόμενη ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται δεκτή όπως έγινε αυτή που έχει τελειώσει. Δηλαδή. δεν μπορεί να αλλάξει πλέον τίποτε. Η ψηφιοποίηση λοιπόν της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας θεωρώ ότι η ψηφοφορία από αυτού έχει ολοκληρωθεί πλέον και είναι δεκτή όπως έγινε. Τώρα, και κανόνες για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροποποιητικός κανονισμός του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με πολλά νούμερα εδώ. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτό. Πάμε στην αρχή λοιπόν, τροπολογία 8. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. 10 και 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 24 υπέρ. Κατά. Α, παρακαλώ, επαλήθευση. 24. Πέρας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια. Δύο, δύο. Σηκώστε καλά τα χέρια. Γιατί τώρα θα χρειάζεται να κάνουμε επαλήθευση. Δύο, επαλήθευση. Πέρασε. Βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, πολύ. Να σηκώνετε καλά τα χέρια για να μπορώ να βλέπω. Τρία και δεκατρία υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχέ. Τώρα χρειάζεται επαλήθευση. Τέσσερα. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν η πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαπέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επτά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαέξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Με ονομαστική κλίση. Αρχίζει. Πέρας. Σαφέστατα εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η επόμενη έκθεση. Να με συμπαθάτε. Εγώ ήμουν. Μα σίγουρα σας θυμίζω τον Σπίτι Γκοντζάλη. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο του κυρίου Μίχαλ Μπόνι. Διαδικτυακή διασυνδεσιμότητα κλπ. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 ε, ναι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έτσι, ναι εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμπεραστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. 61, 61. Με μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν έγινε δεκτή. Να πηγαίνω λίγο πιο σιγά μάλλον, ε για να έχετε και το χρόνο σηκώνετε τα χέρια. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 135. Πέρας. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση πάλι. 136. Πέρας. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση 155. Πέρας. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά επαλήθευση. Επαλήθευση. 175. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές. Με συγχωρείτε, επαλήθευση. 189. 189. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή. 17 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά επαλήθευση. 194. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική βέβαια. Ε. 216 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ κατά επαλήθευση. 226. Πέρασε. Απερίφθη. 2.27 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση και πάλι. 227. 227. Πέρας. Απελήθηκε αυτή. 228 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. 228. 228. Πέρας απεριφθήκε αυτή. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. 230. 230. Πέρας. Απόρριψη. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πολιτισμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πολιτισμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, μεταφορές 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά ε, Παλήθευση 15. 15. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Ας επαληθεύσουμε καλύτερα. 18. Πέρας. Απερίφθη. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α την επαληθεύσουμε και αυτήν. 19. Πέρας. Απερίφθη. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές όχι επαλήθευση Πέρας. Απόρριψη. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κρίση. Αρχίζω. Για το σύνολο της εκθέσεως. Πέρας. Σαφέστατη η πλειοψηφία υπέρ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ δε πολύ όλες και όλους. Εδώ λίγη η ψηφοφορία. Well, uh, I've got some responsibilities in the security of gas supply negotiations now, so I, unfortunately, I should leave. Δυστυχώς πρέπει να φύγω. Και θα ζητήσω από τον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Χένκελ, να αναλάβει στην Προεδρία της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Σπίτι Γκονζάλες. Μεγάλη τιμή να αναλαμβάνω την Προεδρία. Από τον Σπίτι Γκονζάλες στο spider Πάμε για, στη στρατηγική για την Ευρώπη. Διαστημική στρατηγική η οποία θα ενισχύσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, για πολλά χρόνια και βεβαίως είναι ιδιαίτερο σημαντική. Η Επιτροπή Ήτρε έχει κάνει μια δημόσια ακρόαση 10 ε, Νοεμβρίου του 2016 για το θέμα αυτό και έχει κάνει και ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς και την Επίτροπο Βιενκόφσκα και τον κύριο Βέρνερ Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Έχουμε 45 λεπτά για να κάνουμε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην συγγήτρια, την κυρία Κρέλ, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι η συγγήτρια για την έκθεση αυτή Καταρχά θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια πλήρη πρόταση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το διάστημα και νομίζω ότι είναι αυτό ένα πολύ καλό μήνυμα γιατί όντω η πολιτική για το διάστημα για πολλού. Ε, ε, σημαίνει κάτι πολύ εξωγήινο, αλλά παρόλα αυτά επηρεάζει ιδιαίτερο σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη, τις κοινωνικές διαδικασίες και γι' αυτό θεωρώ ότι ως Κοινοβούλιο και εμείς πρέπει να λάβουμε θέση. Κάτι που κάνουμε μέσω της εκθεσής ε, μου. Ευχαριστώ και τους κοιόδες συζητητές μου ε, για την καλή συνεργασία. Νομίζω ότι είναι καλή λοιπόν αυτή η δυνατότητα για να θέσουμε τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε και το Γαλιλαίο και το Κοπέρνικους, ε, το οποίο τα οποία ούτως ή άλλως θέτουν κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες. Βεβαίως αυτές πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται ε, και βεβαίως ε, να, να τις οικειοποιηθούν τα κράτη-μέλη. γιατί βεβαίως πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα ε, κονδύλια για να μπορούμε να ανανεώσουμε τον στόλο μας και την γενιά των συσκευών που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό, το θέμα ε, των ε, διαστημικών απορριμμάτων. Η υπηρεσία προετοιμάζει πάρα πολλά ως προς αυτό και ενεργώς δουλεύει πάνω στο θέμα αυτό και επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία δεν είναι θεσμικό ευρωπαϊκό όργανο, είναι η... μια υπηρεσία ευρωπαϊκών χωρών αλλά και μη ευρωπαϊκών χωρών που όλα μαζί συνεργάζονται και νομίζω ότι ακριβώς η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΖΑ είναι πραγματικά πολύ καλή και θα πρέπει να εξελιχθεί έτσι ε, περαιτέρω για να μπορέσουμε να ε, διαχειριστούμε από κοινού όσα προκύπτουν. Επίσης, σημαντική πρόκληση είναι τα ερωτήματα των, ε, του κυβερνοχώρου και αυτό είναι ούτως ή άλλως ένα κομμάτι της υποβληθής σας έκθεσης. Τώρα για το downstream της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας διαστήματος είναι πολύ σημαντικός ο τομέας αυτός βιομηχανίας για την οικονομία και θα πρέπει όντως να δούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έτσι ώστε να τους διευκολύνουμε τη ζωή να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα και για τα επιχειρησιακά μοντέλα το Γαλιλαίο και το Κοπέρνικους και βεβαίως να τους βοηθήσουμε για την πρόσβαση σε τέτοιου είδους ιδέες και προγράμματα. Χρειαζόμαστε μεταξύ άλλων μια πιο απλοποιημένη διαδικασία πρόσβασης σε δεδομένα, αλλά κυρίως θα πρέπει να κατανοήσουμε και να καταφέρουμε τα συστήματα λήψη ε, να είναι συμβατά με το σύστημα του Γαλιλαίου. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν κάποια πρότυπα. βεβαίω, η βιομηχανία έχει το δικό τη συμφέρον προ αυτό, αλλά όταν δεν αρκεί το ιδιωτικό συμφέρον, η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι εμείς να ενδιαφερθούμε περισσότερο έτσι ώστε να πλαισιώσουμε τις προσπάθειες αυτές με νομοθεσία. Βεβαίω θα πρέπει πρώτα η βιομηχανία να δει τι μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά νομίζω ότι και εμείς, έστω συντηρητικά στην αρχή, θα πρέπει να παρέμβουμε. Κατά την άποψή μου, η περιφερειακή διάσταση επίσης πρέπει να τονιστεί, γιατί ακριβώς στις περιφέρειες υπάρχουν πολλές δυνατότητες εφαρμογής και χρήσης, οι οποίες συχνά δεν, είναι, δεν έχουν γίνει κατανοητές από τις περιφέρειες. Ας πούμε στην πολιτική συνοχή, στην ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κίνητρα για τον τομέα αυτό, ώστε να δραστηριοποιηθούν ακόμη περισσότεροι upstream τώρα της, ε, βιομηχανικής, ε, της ε, βιομηχανίας. Θα πρέπει να δούμε το επίπεδο προστασίας, θα πρέπει να προστατέψουμε από αθέμητο ανταγωνισμό τρίτων χωρών. Ο δίκαιος, ο θεμητός ανταγωνισμός βοηθά να ενισχυθεί ο τομέας και θα πρέπει να μην τον επηρεάζουμε με οποιοδήποτε είδος περιοριστικές εγγύησεις. Επίσης, ο ρόλος των δορυφόρων για τις τηλεπικοινωνίες. Πολύ σημαντικό θέμα για τη συνδεσιμότητα και την κάλυψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση με ε, ίντερνετ υψηλή ταχύτητα, όχι μόνο για τις απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και για τις ε, πιο ε, υποβαθμισμένες περιοχές. Εκεί λοιπόν πρέπει η διαθεσιμότητα να υπάρχει με τις συγκεκριμένες συχνότητες, για τον προπολογισμό τώρα θέλω να πω δύο πράγματα. Ξέρουμε ότι οι δραστηριότητε ε, στο διάστημα αυξάνονται κυρίως λόγω και της αύξησης της ψηφιοποίησης και βεβαίως αυτό είναι αρκετά κοστοβόρο. Είναι βεβαίως ε, σημαντική η προστιθέμενη αξία του κλάδου αυτού, γι' αυτό και εμείς ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχουμε τον απαραίτητο, για να ζητήσουμε τον απαραίτητο προπολογισμό για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να καταστήσουμε σαφές ότι εδώ θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τα οικονομικά. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι σαφής η διακυβέρνηση, η διαχείριση. Γι' αυτό εγώ ζητώ την, από την ΕΖΑ και από, την, ε, ε, το Παγκόσμιο Διορφορικό Σύστημα Πλοήγησης και από την Κομισιόν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο έτσι ώστε να προχωρήσουμε ως προς το θέμα της διαχείρισης. Τέλος, ασφάλεια στο διάστημα που συνδέεται ε, πολύ στενά με όλα αυτά. Ε, πρέπει να είμαστε τυπικοί με τα προγραμματά μα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κυρίω ό,τι αφορά την διάσταση τη ασφάλεια. Συζητούμε για, ένα, για μια πολιτική ε, ευρωπαϊκή Άμυνα και ασφάλεια, οπότε πρέπει να προσέξουμε τα προγράμματα για το διάστημα να τα εντάξουμε και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Κρέλ. Πήρατε λίγο παραπάνω από 6 λεπτά. Έχουμε τώρα δύο λεπτά για τους εισηγητές. Η κυρία Σαντέρ θα ε, αντικαταστήσει την κυρία Γκροστέτ, την Σκιώδη. Η κυρία Σαντέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα όντω να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματο τη κυρία Γκροστέτε που χρειάστηκε να μείνει στο Παρίσι για μια πολιτική ε, συνεδρίαση και θα σα διαβάσω το κείμενο που είχε προετοιμάσει. Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτη, την κυρία Κρέλ για το σχέδιο έκθεση που αποτελεί μια στέρεη ε, βάση εργασία και που συμπεριλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία. Είναι πρώτη φορά που έχουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση για μια πραγματική ε, ε διαστημική και στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ένα και περισσότεροι τομεί ε, ε, ε, θίγονται από τι πρόοδους, θετικά ή αρνητικά από τις πρόοδους της διαστημικής τεχνολογίας. Έχουμε να κάνουμε την αλληλεία, τη γεωργία, την άμυνα, τη διαχείριση συνόρων και άλλους τομείς. Η μείωση του ψηφιακού της διαστημικη που έχει δημιουργηθεί χάρη στους δορυφόρους θα εξυπηρετήσει όλους τους τομείς και αλλου τομει η μειωση του ψηφιακου ρηγματο που εχει δημιουργηθει χαρη στου δορυφορου θα εξυπηρετησει ολου του τομει και ολου κόσμο, στους συμπολίτες. Ο διαστημικός τομέας είναι πολύ στρατηγικός και ευαίσθητος, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει δραστήριο ρόλο για να εγγυηθεί ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα για την Ευρώπη, ιδίω στο, στα θέσεις διεθνέ πλαίσιο που γνωρίζουμε. Γι' αυτό η δημόσια στήριξη πρέπει να είναι ισχυρή, γιατί η διαστημική βιομηχανία δεν μπορεί να μείνει μόνη έναντι του διεθνού ανταγωνισμού. Πρέπει να το επιτρέψουμε να είναι ανταγωνιστική. Πρέπει επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την ανάπτυξη των δικών τη εκτοξευτών όπω το Αριάν και το Βέγγα, ε, το συμφέρον τη ύπαρξη. Ε, ευρωπαϊκών εκτοξευτών είναι σαφή ανεξαρτησία και βιομηχανικό ατού στην Ευρώπη με δημιουργία 40.000 θέσεων απασχόλησης. Ε, το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να είναι σωστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρχει αποδοτικό αυτών των εκτοξευτών. Επίσης, στήριξη στις υποδομές όπως ε, το διαστημικό λιμάνι του Κουρού που είναι στρατηγικό σημείο για την εκτόξευση διορυφόρων είναι απαραίτητη. Τέλος, χρειάζεται να υποστηρίξουμε αυτήν την πτυχή ε, ε, που προηγείται αν θέλουμε να στηρίξουμε και την ανάπτυξη κατόπιν της εκτόξευσης. Η ανάπτυξη λοιπόν γενικά θα πρέπει να ευνοηθεί στο διαστημικό τομέα, μικρομεσαίες να υποφεληθούν από αυτή την προσπάθεια και να διευκολυνθεί και η πρόσβαση στα διαστημικά στοιχεία, πράγμα που δεν συμβαίνει πολύ ε, σήμερα σε σχέση με την εκπομπέ τις εκπομπές του άνθρακα, στηρίζω την πρόταση τη της Θα θέλω να ε, διευρύνω σε όλου του ρήπου. Ε, που, έχουν, ε, που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα μπορούσαμε ας πούμε, να το διευρύνουμε και στο μεθάνιο. Οι προπολογισμοί για το διαστημικό μας πρόγραμμα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι γιατί σε ολόκληρο τον κόσμο αυξάνονται οι σχετικοί προπολογισμοί και θα πρέπει να έχουμε τα μέσα για τέτοια διαστημικά προγράμματα όπως το Γαλιλαίο, Κοπέρνικος ε, και ούτω καθεξής. Διαστημικό τομέα είναι επένδυση στο μέλλον και δεν θα το μετανιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν επενδύσει στο διάστημα. Ευχαριστώ. η κυρία του Κοζανό, ο κύριος, συγγνώμη, Κοζανόσκη. Καταρχάς, να συγχαρώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Έχουμε συνεργαστεί και για το για τον φάκελο αυτό και την αγορά και χαίρομαι που τα συνδέει η συγκέντρια. Έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την ε, τεχνολογία στα πλαίσια του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικου. Δυστυχώ η Κομισιόν εντωμεταξύ έχει υποβάλει νέε προτάσει, οι οποίε δεν έχουν ε, περάσει από αυτό το space check που, που λέμε. Ε, ας πούμε για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Και κάποιες άλλες πτυχές που αναφέρει η κυρία ε, Κρέλ και που συνδέονται με το φάκελο αυτό. Μιλούμε για τι ε, συνδέσει μέσω δορυφόρου υψηλή ταχύτητα. Βεβαίω είναι καλό, αλλά πρέπει να είναι συμβατό με τα δίκτυα 5G και θα πρέπει να καλύψει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω είναι καλό αυτό και είναι πολύ σημαντική πτυχή. Επίση, στην έκθεση μιλούμε για την ενδιάμεση θεώρηση του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικου και αυτό είναι καλό. Και είμαι πεπισμένο ότι θα υπάρξει ε, συνέργεια και θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε την ασφάλεια του Κοπέρνικου. Η κυρία Κρέλ δικαίω μιλά για τις ε, τρίτε χώρε στην εκθεσή τη. Εδώ θέλω ξανά να κάνω έκκληση γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα του, της Μεγάλης Βρετανίας που είναι ο πιο σημαντικός εταίρος μας στην πολιτική του διαστήματος. Και επίσης το GovSatcom, η σχετική πρωτοβουλία και η υπηρεσία SST. Η ομάδα μας βρίσκεται περίπου ανάμεσα στην μάλλον προτιμά τις, ε, την, ε, τη διακρατική συνεργασία παρά την ε, δημιουργία νέων προγραμμάτων. Οπότε ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ που τηρέστηκε το χρόνο σας. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Κρέλ για την πολύ καλή δουλειά της και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα μίλησε με, τους, ε, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι πολύ καλή η αρχή αυτή. το σχέδιο έκθεση είναι ισόρροπο, που και καταγράφει τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε όντως να έχουμε επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική για το διάστημα. Ε, πρέπει να έχουμε έναν υγιή τομέα για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική και αυτό θέλω να τονίσουμε στην έκθεση. Καταρχάς την αύξηση στις επενδύσεις, στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, και επίσης το πρόγραμμα 9 και το, το πρόγραμμα πλαίσιο 9 και η γραμμή του προπολογισμού. Ε, το, η πολιτική είναι πολύ σημαντική γιατί μιλούμε για τις τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρων, υψηλή ταχύτητα, ίντερνετ υψηλής ταχύτητας, το, τα small set launchers. Αν θέλουμε να είμαστε λοιπόν πρωτοπόροι, θα πρέπει να ενισχύσουμε πρώτα την έρευνα. Δεύτερον, που σχετίζεται με αυτό, είναι ότι πρέπει να υποστηρίζουμε αυτά που λέμε με πράξεις, με κονδύλια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε γιατί αγοράζουμε δεδομένα εκτός Ευρώπης και γιατί δεν χρησιμοποιούμε τηλέφωνα που να ε, είναι συμβατά με τον Γαλιλαίο. Κυρίως εδώ οι εργαζόμενοι πούμε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από αυτούς. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει, και το είπε και η κυρία Κραλίδη, ε, με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Νομίζω ότι χρειάζεται καλύτερα ε, πρότυπα γιατί η υποδομή μας που είναι ψηφιακή για το διάστημα είναι πραγματικά πάρα πολύ ευαίσθητη. Οπότε η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες ε, υπηρεσίες έχουν, έχουν δυνατότητα αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων. Και τέλος η στρατηγική επικοινωνία. Το είπαν και κάποιοι άλλοι ομιλητές αν θέλουμε να επενδύσουμε στο διάστημα, χρειαζόμαστε δημοκρατική υποστήριξη ως προς αυτό. Και κατά την άποψή μου, η στρατηγική για την επικοινωνία θα πρέπει να έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι να αυξήσουμε την επιστοποίηση του κοινού. Το κοινό πρέπει να κατανοήσει τι ακριβώς έχει να λαμβάνει από αυτή τη διαδικασία, ότι όντω αυτή η πολιτική είναι κομμάτι της καθημερινής του ζωής. Η επικοινωνία λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο ε, προσγειωμένη. Η εκπαίδευση επίση στα σχολεία πρέπει να εμπνεύσουμε τα μικρά παιδιά να γίνουν οι μελλοντικοί επιστήμονες, οι μελλοντικοί αστροναύτε. Τώρα χρειαζόμαστε μονίμως άτομα εκτός Ευρώπης να δουλέψουν για τον δικό μας ευρωπαϊκό τομέα του διαστήματος. Και ο τελευταίος πυλώνας, και επίση αναφέρθηκε, είναι οι επιχειρηματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες των προγραμμάτων που έχουμε. Πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Κοπέρνικου δωρεάν, ας πούμε. Αυτοί λοιπόν οι τρεις πυλώνες νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ε, αυτοί που θα πρέπει να τονιστούν στην ε, στρατηγική επικοινωνία και βεβαίω ε, με χαρά θα συνεργαστώ με του κοιόδε και με την κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, ο κύριο Κούλιτσεκ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε. Έχω ορισμένα σχόλια. Με την κυρία Κρέλ οι εμπειρίες που έχω από τη συνεργασία μαζί της είναι εξαιρετικές. Οι συζητήσεις και με άλλους και ηγητές είναι πραγματικά ε, Ελπίζω να συνεχιστεί στο μέλλον. Αυτό το space check είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Οφείλουμε να επιμείνουμε στην πραγματική του εφαρμογή. Αφενός. Αφετέρου, οι διασυνδέσεις υψηλής ταχύτητας που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Πολύ σημαντική επίσης η έρευνα και η ανάπτυξη. Για τις μεταφορές, που οι μεταφορές μέχρι τώρα δεν συζητήθηκαν. Και όμως ανοίγεται εδώ μια τεράστια δυνατότητα για πρόοδο και σε συστήματα διοδίων. Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις που αναφέρονται στα συστήματα πράξης διοδίων. Αν αφήσουμε τις παλές τεχνολογίες μικροκυμάτων, τότε βλέπουμε ότι ο Γαλιλαίος μπορεί να μας βοηθήσει να εισπράττουμε διόδια με ενίο τρόπο, αν και θα υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες μέλη, εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας τέτοιες τεχνολογίες, θα πρέπει να επιλέξουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Και για την νεολαία έχουμε εμεί στην Τσεχική Δημοκρατία από καιρού ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ε, σημαντικό και επιτυχημένο πρόγραμμα το οποίο ε, προκαλεί το ενδιαφέρον των νέων για το διάστημα. Και φέρει και το όνομα του Γκαγκάριν, του παλαιού αστροναύτου. Ευχαριστώ και ο Κύριο Σαφχάουζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα ό,τι έχει σχέση με το διάστημα είναι αρμοδιότητας των κατών και ιδίως της Γαλλίας. Άλλωστε υπάρχει και μια διακυβερνητική οργάνωση, η ΕΣΑ, που πράγματι πρέπει να υποστηριχτεί. Η Ευρώπη θα αναζητήσει τη θέση της στην εναρμόνιση, στη χρηματοδότηση της διακυβερνητικής συνεργασίας και πάντως όχι για να δημιουργήσει ένα καινούριο γραφειοκρατικό οργανισμό ή όπως είδαμε και με τον Γαλιλαίο, προγράμματα τα οποία μετά η Ευρώπη δεν μπορεί να διαχειριστεί. Ούτε και είναι ικανή να τηρήσει τον ίδιο τον οδικό χάρτη τον οποίο απεφάσισε. Ιδίως να προσέξουμε το πρόβλημα της ασφάλειας και της άμυνας που πάλι είναι ζήτημα αρμοδιότητας των χωρών μελών. Και κάθε φορά που παρεμβαίνει η Ευρώπη το κάνει με πλήρη ανικανότητα δράσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη απαραίτητα την κυριαρχία των χωρών μελών, όπου πάλι εκεί δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Ευρώπη. Εγώ έχω εργαστεί ο ίδιος στο πρόγραμμα μικροδορυφόρων και των οχημάτων που τα μεταφέρουν αυτά τα πράγματα στο διάστημα. Πάλι εκεί διόλου δεν έχει ικανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμαστεί για το μέλλον. Ό,τι αφορά την διακυβερνητική συνεργασία λειτουργεί καλά, ό,τι αφορά τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα δεν τα καταφέρει να λειτουργήσει. Άρα, να υποστηρίξετε τον ΕΑΣΑ και φτάνει. Ευχαριστώ αγαπητέ Σαφχάουζερ, εισηγητής ογνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών κυρία Μέισνερ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ο Κόχλησεκ μίλησε πριν για τη διασύνδεση με τις μεταφορές. Και η στρατηγική αυτή έχει πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις μεταφορές και για την ίσπαση διοδίων αλλά και γενικότερα για την ψηφιοποίηση των μεταφορών που θα οδηγήσει σε λιγότερα σημεία εχμή στην κυκλοφορία και ούτω καθεξής. Θα χρειαζόμαστε αυτά τα πράγματα. Εκτός όμως από τον τομέα των μεταφορών, δώστε μου ένα λεπτό για να σας πω για κάτι άλλο το οποίο συχνά λησμονείται η πολιτική της θάλασσας. Υπάρχει μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλίας, αλλά εκεί μιλάει μονάχα για την παράνομη αλία. Βεβαίως ο δορυφόρος δεν μπορεί να κοιτάξει μέσα από το νερό και μέχρι το βυθό της θάλασσας. Μπορεί να δει όμως τι γίνεται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, να παρακολουθεί ε, παράνομες δραστηριότητες, ε, ρήπανση του περιβάλλοντος, παρανομιαλία, άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. έρευνες και μελέτες στην επιφάνεια της θάλασσας που μπορεί να επιτρέψει λοιπόν πολύ ε, την άσκηση της πολιτικής αυτής και για την καθαριότητα των ωκεανών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Χένκελ, ο κύριος Ρούιμπικ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Με ενδιαφέρει η μελλοντική στρατηγική τι θα κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον για να οργανωθούμε καλύτερα στον χώρο αυτό. Η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών χρειάζεται βελτίωση. Δεν είναι μόνο ο GNSS, ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος και η ΕΣΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Και αυτή φύγεται εδώ. Τι γίνεται και με την ΕΝΙΣΑ. Εδώ μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα με συνεργασία. Και άλλοι οργανισμοί αφορώνται εδώ. Χρειάζεται μια στρατηγική ώστε να ενισχυθούν και επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας μπορεί να συμβάλλει ώστε στον τομέα αυτό έγκαιρα να ισχύσουν ψηφιακές προδιαγραφές, κάτι που για την ευρωπαϊκή οικονομία θα σημαίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Κυρίως η εφαρμογή σε πραγματική κλίμακα θα παίξει σημαντικό ρόλο, διότι έτσι θα προκύψουν παγκόσμια πρότυπα. Με ενδιαφέρει επίσης και αυτά με ενδιαφέρουν αυτά τα κλάστερ, αυτές οι, ε, αυτά τα κλάστερ της ε, διανοητικής ιδιοκτησίας Πώς οργανώνονται αυτά. Πώς έχουν προχωρήσει τα πρότυπα εκεί που θα ισχύσουν για τα εγχειρήματα αυτά στο μέλλον και ιδίως ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Και βεβαίως και η επικοινωνία μεταξύ των διαφορών οργανισμών, επαναλαμβάνω όπως είπα στην αρχή, ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί. Η κυρία Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και από μένα προς την εισηγήτρια για τη θαυμάσια έκθεση που έχει συντάξει. Έχει βέβαια η στρατηγική διαστήματος κάτι να προσθέσει στο έργο που έχει γίνει ως τώρα. Έρχομαι όμως ιδίως σε αυτά που λέχθηκαν για τα απορρίμματα στο διάστημα, που για μας έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θέλουμε να προχωρήσουν κάποια προγράμματα. Και η εξερεύνηση του διαστήματος, που κάπως ακροθυγώς το περνάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμά της, αλλά και για τον περιορισμένο προϋπολογισμό με τις υφιστάμενες δυνατότητες χρηματοδότησης για τα μη στατιωτικά προγράμματα. Εάν δούμε όμως στατιωτικά προγράμματα, τότε χρειάζονται και άλλα κονδύλια από τις χώρες μέλη. Ας το έχουμε σαφώς υπόψη λοιπόν αυτό στην εργασία μας. Η στατική επικοινωνιών, σημαντικό για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, αλλά και ως έμπνευση για την επόμενη, και τις επόμενες γενναίες Και τέλος, εγώ θα ήθελα πολύ το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει ενεργό μέσα στην ε, ε, πορεία αυτή. Βεβαίω επωφελείται η χώρα μου, αλλά έχει και σημαντικό ρόλο να παίξει στο διάστημα ο πρόεδρος Χένκελ. Ας θυμηθούμε ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το διάστημα δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην Ευρώπη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την συνεργασία με την Ελβετία και βεβαίω και μετά και από τη Βρετανική έξοδο και με την Βρετανία. Η κυρία Μάισνερ νομίζω έδωσε ένα καλό παράδειγμα της σφαιρικότητας του ζητήματος. Ο δε κύριος Ρούμπικ μίλησε επίσης για παγκόσμια ισχύω πρότυπα. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεχίσουμε την συνεργασία αυτή και να την βελτιώσουμε όλες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Κίνα και με τη Ρωσία και με τις Ινδίες και με την Ιαπωνία και με άλλες χώρες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο διάστημα. Ευχαριστώ. Έλερα. Συγχαίρω ειλικρινώς την εισηγήτρια. Πολύ ουσιώδης η εκθεσή της. Και ευχαριστώ επίσης που και το θέμα ότι θέλουμε ένα καινούριο αμυντικό πρόγραμμα, γιατί μέχρι τώρα η διαστημική στρατηγική προχωρεί σε μια τεχνητή διάκριση και τη διατηρεί ανάμεσα σε στρατιωτική και μη στρατιωτική εφαρμογή στο διάστημα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε τώρα αυτό. Μακροπρόθεσμα δεν θα μπορέσει να επιζήσει η Ευρωπαϊκή Διαστημική στατική χωρίς στρατιωτική πτυχή. Είτε διεθνώς, είτε δίνονται σε μη στρατιωτικέ εφαρμογέ πάρα πολύ υψηλέ κρατικέ χρηματοδοτήσει όπω στην Νότια ανατολικη Ασία, είτε συμβαδίζουν με τη στρατιωτική εφαρμογή. Αυτό χρειάζεται λοιπόν να ενταχθεί περισσότερο στην προσπάθεια αυτή. Και στον αμυντικό προγραμματισμό πρέπει να δούμε να δούμε, να μην είναι απλά ένα πρόγραμμα κατανομής κονδυλίων, αλλά να δούμε ποιοι τομείς είναι εκείνοι που πρέπει να ενισχυθούν ευρωπαϊκά. Γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ της ιδέας να ανοίξει η συζήτηση για το ζήτημα ενός νέου στρατιωτικού ερευνητικού προγράμματος με επίκεντρο το διάστημα. Να αποτελέσει αυτό δηλαδή ένα πυλώνα στον οποίο θα στηριχτεί η μελλοντική διαστημική δραστηριοποίηση της Ένωσης. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για προστασία συνόρων κλπ. κλπ εάν δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά, να, να, να υπάρχει μια οπτική εικόνα όλων αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν πρόκειται για την στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Πρόκειται για μια λογική προσπάθεια διασύνδεσης παράλληλων προγραμμάτων κ. Ντασίλβα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Commission... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή θα ήθελε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια την κυρία Κρέλ ε, η έκθεση που συνέταξε και που μόλις μελετήσαμε είναι πολύ καλή και η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Κρέλλα εντοπίζει σωστά τις προτεραιότητες που έχουμε εμείς ε, θέσει επιτάπητος, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιοι είναι οι κίνδυνοι του, ε, της στρατηγικής αυτής. είναι σαφές ότι Αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε είναι να φέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες τα πρώτα μηνύματα για το τι θα ωφεληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι κοινοτικές πολιτικές. Αυτή ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα και χαιρόμαστε που βλέπουμε να υπάρχει συνένεση με αυτή μας την ε, ε, την ε, πρόθεση. Είναι σημαντικό λοιπόν να φτιάξουμε την, ε, μια τέτοια στρατηγική και να την εφαρμόσουμε καθώς και σημαντικές είναι οι ε, συνέπειες ε, της εφαρμογής αυτής στο μέλλον για το σύνολο των κοινοτικών πολιτικών. Τα μέσα τα οποία θα είναι διαθέσιμα πρέπει να, ε, να είναι σε ισορροπία με αυτή την διαστημική πολιτική. Θα πρέπει να σκεφτούμε πως υπάρχουν πολλοί θεσμοί που είναι αρμόδιοι για την διαστημική ε, πολιτική. Πρώτα απ' όλα το Ευρωκοινοβούλιο, μετά το Συμβούλιο, μετά τα κρατημέλη, μετά ο Ευρωπαϊκός ε, Διαστημικός Οργανισμός, ε, η, ο Οργανισμός της Πράγας και άρα είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ο διάλογος με όλους τους θεσμούς και άρα και με την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία ένταξης, όπως το κάναμε και σε αυτή τη στρατηγική, για να μπορέσουμε πραγματικά να εντοπίσουμε τις προτεραιότητες και να τις διευκρινίσουμε, να διευκρινίσουμε το ρόλο του καθενός Κομισιόν, Κράτο, Μέλη, Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός, όλων των θεσμών λοιπόν, έτσι ώστε εν τέλει να μπορούμε να είμαστε αποδοτικοί και να φέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες τα ωφέλη και να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσουμε τον σημαντικό ρόλο της διεθνικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, συνοψίζοντας η θέση της Κομισιόν σε αυτό το στάδιο είναι ε, η εξή. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα ε, που θα προκύψουν στη διάρκεια της συζήτηση, αλλά η έκθεση αυτή που εκπώνησε η κυρία Κρέλ για την Επιτροπή είναι καλή έκθεση και εντοπίζει σωστά τις προτεραιότητες της Ένωσης, ε, τα, τις προκλήσεις επίσης, τους κινδύνους και δεν θα πρέπει να κρύβουμε και να μασάμε τα λόγια μας και τη κρίσιμα στοιχεία των όσων έχουμε πράξει μέχρι στιγμής και των όσων προτιθέμεθα να κάνουμε στο μέλλον και για τα οποία και κλείνω θα πρέπει πραγματικά να έχουμε μια υποστήριξη ευρεία για να μπορέσουμε να έχουμε το... τα μέσα στη διαθεσή μας και να τα αποκριθούμε στις προκλήσεις. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας επένεσαν πάρα πολύ όλοι οι συνάδελφοι, άρα θα σας αφήσω κυρία Κρέλ λίγο περισσότερο χρόνο για να μπορέσετε να μιλήσετε. Δεν θα ακρηγορήσω πλέον, όχι. Με μία εξαίρεση μου φάνηκαν όλα πολύ ομοιογενή τα σχόλιά σας. Με μία εξαίρεση επαναλαμβάνω. Θα ήμουν ευγνώμων εάν είναι δυνατόν τα όσα συμπληρωματικά μνημονεύσατε να λάβουν τη μορφή τροπολογιών. Βεβαίως γνωρίζετε ότι έχω περιορισμό στα όσα μπορώ να συγγράψω ε, εκ των κανονισμών του Κοινοβουλίου. Αναμένω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τι προσθήκε που ενδεχομένω θα θέλετε να επιφέρετε. Ευχαριστώ. Προθεσμία καταθέσει τροπολογίων, λέει ο Πρόεδρο, είναι η 26η Απριλίου. Άρα δεν σα μένει πολύ καιρό. Το τελευταίο τώρα θέμα τη σημερινή ημερησία διατάξεω είναι η αξιολόγηση του προγράμματος, της υλοποίησης του προγράμματο ορίζοντα 2020 με ναι, γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο. Συνολικά έχουμε μαζέψει 372 τροπολογίες. Ελπίζω οι σκληρότητες συγητές να συμφωνήσουν γρήγορα να περιορίσουν τις τροπολογίες αυτές, να τις ε, περιλάβουν στις συμβαστικές για να απηχούνται καλύτερα οι απόψεις όλων των ενδιαφέρων μερών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας μένουν 45 λεπτά για τη συζήτηση αυτή. διότι χάσαμε κάποιο χρόνο και με την συζήτηση περί της ψηφοφορίας, όσο θα θυμάστε. Να δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή κύριο Ρούες. Κυρία Λουίς, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως θα τα πω λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Προβλήθηκαν 372 τροπολογίες και η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι δυνατόν να φτάσουμε σε συμφωνία γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών αυτών στόχο έχει να βελτιώσει το κείμενο και θα μπορέσουμε νομίζω έτσι να φτάσουμε σε συμφωνία. Δεν χρειάζεται να ξαναμιλήσω για τα θέματα. Υπάρχουν ε, θέματα. Θα προχωρήσω λοιπόν κατευθείαν σε δύο σημεία όπου πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε πιο διαφορετικές απόψεις και όπου νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση από πλευράς της επιστημονικής κοινότητας και ε, περισσότερες αντιδράσεις ακούσαμε ότι μεγάλη βιομηχανία. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα όσον αφορά την αξιολόγηση. Εξ αρχής θέλω να πω ότι η αριστεία που κατά την γνώμη μου θα πρέπει να, ε, να συνεχιστεί γιατί είναι ο βασικός άξονας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα γεωγραφικά κριτήρια αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε αναφέρει και θέλω να πω ότι έχουμε και χρειαζόμαστε περισσότερη ρηστή από αυτή που χρειαζόμαστε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε λοιπόν τους μηχανισμούς και τους τρόπους ώστε να δημιουργηθούν περισσότερα ακόμα κέντρα αριστεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μιλήσει και για κάποια μέτρα όπως η καλύτερη μισθή για τους ερευνητές και ούτω καθεξής. Και όσον αφορά το φύλλο, ε, παραπέμπουμε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2015 που λέμε για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και γι' αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε το θέμα της απουσίασε των γυναικών. Θα πρέπει βεβαίω να βελτιωθεί και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά πιστεύω ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο από την άποψη την οικονομική, την άμεση και άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε πώς, να μας προβληματίσει πώς θα αναπτυχθεί και κοινωνικά η αριστεία. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά τα λίγα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Η μεγάλη βιομηχανία βεβαίως ε, παίζει ρόλο όταν έχουμε project με μεγάλη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και άρα λοιπόν θα πρέπει να καλέσουμε περισσότερο για συμμετοχή ε, σε αυτό το 3% του ΑΕΠ. Χρειάζεται να συμμετέχει κατά 65% ο ιδιωτικός τομέας, η μεγάλη βιομηχανία, η βαριά μας βιομηχανία και πρέπει να καταβάλουμε μια παραπανήσια προσπάθεια ώστε αυτό να το καταφέρουμε και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Φυσικά είμαι διαθέσιμη για συνεργασία με όλους και θα δώσουμε τώρα το βήμα στις διάφορες ομάδες που κατέθεσαν τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ κυρία Ρουίθ και τώρα εξ ονόματος του ΕΛΚ κυρία Κουτρίτσκα. Δύο λεπτά. Να σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, όντως, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε συμβιβαστικές. Εμείς, για παράδειγμα, προτείναμε 170 τροπολογίες ε, ε, Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να θεσπιστεί ένας προπολογισμό για, την, ε, για τις ε, επιστήμες, για την έρευνα. Ε, το Κοινοβούλιο δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να πάρει όλα αυτά που ζητάει από την Κομισιόν. Και... Εδώ λοιπόν έχουμε και θέλουμε να φτιάξουμε στη συμβεβαστική, να διατηρήσουμε τη σημερινή δομή του προγράμματος με κάποιες απλοποιήσεις. Πιστεύω πως και ε, ότι θα μπορέσουμε λοιπόν να φτάσουμε στη συμβαστική λύση. Θα πρέπει να σκεφτούμε τις κοινωνικές προκλήσεις και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες συνδέσεις ανάμεσα στα προγράμματα και συνεργασίες. Προβλέπουμε και την δημόσια στήριξη, αλλά και δείκτες επιτυχίας. θα θέλαμε δεν να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στη βιομηχανία και του, τους επιστήμονες. Να υπάρχουν ΣΔΙΤ, οι μικρομεσαίες να μπορέσουν να συμμετέχουν σε project και να σκεφτούμε επίσης και κίνητρα για τη βιομηχανία. Στηρίζουμε δε την ανοιχτή πρόσβαση γιατί δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε κάτι στην βιομηχανία. Αυτή ε, καθοδηγείται από τον ανταγωνισμό. Επίσης θεωρούμε πως η άμυνα θα πρέπει να είναι έξω από το πρόγραμμα πλαίσιο. Το 44,7% θα πρέπει να ε, προορίζεται για τα νέα κράτη-μέλη από τα κονδύλια. Και τέλος, το πιο σημαντικό μας κριτήριο θα πρέπει να είναι η επιστημονική αριστεία. ECR, ε η κυρία Φαν Μπόσελτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ήδη συζητήσει μια φο... κάποιες φορές τον ορίζοντα 2020 και θα το ξανασυζητήσουμε στο μέλλον. Εγώ είμαι ικανοποιημένη από την εργασία της εισηγήτριας. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες, ωστόσο, αλλά πρόκειται περισσότερο για ε, εμβάθυνση στα όσα ήδη έχει κάνει η εισηγήτρια. Τώρα θέλω να πω ε, τέσσερα σημεία που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, απλοποίηση διοικητική των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ε, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν ήδη έχει αρχίσει μια τέτοια προσπάθεια. Όμως μέχρι τώρα η απλοποίηση έχει γίνει περισσότερο προς της ίδιας της Κομισιόν, ενώ θα έπρεπε να ε, ε, επιμείνουμε στο να ωφεληθούν οι επιχειρηματίες. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει περισσότερος προσανατολισμός στις επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες, ε, αλλά όχι μόνο, αλλά να υπάρχει ίσως ένα χαμηλότερο επιτόκιο ε, για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτές ε, τις δράσεις. Ο το ορίζον 2000 θα πρέπει να θεωρηθεί ως διευκόλυνση για την ανάπτυξη. Τρίτον, δύο φάσεις ε, έχουμε για την εφαρμογή. Αυτό είναι χρήσιμο όργανο και εργαλείο μάλλον σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία επιλογής. Όμως, πιστεύω ότι ότι χρειάζεται πιο συγκεκριμένος καθορισμός στις πρώτες φάσεις και πιο αυστηρά κριτήρια για να μην περάσουν τόσοι πολλοί ε, ενδιαφερόμενοι στη δεύτερη φάση. Τελευταία παρατήρηση να μετατραπούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα ευρήματα της ευρωπαϊκής έρευνας ε, που μέχρι στιγμής παραμένει σε επιστημονικό επίπεδο, δηλαδή στα, στα πανεπιστήμια. Πρέπει να μπορέσουμε να καταφέρουμε να ε, εφαρμοστούν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών. Να σκεφτούμε και το πλαίσιο των ε, επισφαλών κεφαλαίων, venture capitals, και να φτιάξουμε και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Καινοτομίας. Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία στην εισηγήτρια εύχομαι και καλή δουλειά για τις συμβιβαστικές. Ε, ε, ε, είμαι βέβαιη ότι θα πετύχουμε καλό αποτέλεσμα και να πούμε έτσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι αναμένει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Horizon 2020 και από το μελλοντικό ερευνητικό μας πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίρινγκ. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να πω ότι με εντυπωσιάζει ο ρυθμός των ε, τροπολογιών. Σχεδόν 400 ε, διαπιστώνω ότι υπάρχει μέγα ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της έρευνας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που είναι θετικό. Ταυτόχρονα είδα ότι αυτές οι 400 τροπολογίες είναι ενδιαφέρουσε. Υπάρχει δηλαδή υλικό και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε. Εγώ μαζί με του φιλελεύθερου συναδέλφου, έχω υποβάλει τροπολογίες και υπογραμμίζω πως στόχο είναι να βελτιωθεί περισσότερο αυτή η έκθεση βασικό θέμα είναι ότι αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, όχι μόνο λόγω μεγαλύτερου προϋπολογισμού, αλλά και λόγω του ότι επικεντρώνεται στην διασυνοριακή συνεργασία και αυτά είναι πράγματα που τα θεωρούν σημαντικά όλοι οι φορείς. Τα κριτήρια αριστείας λοιπόν θα πρέπει να μαζί με αυτά τα κριτήρια να αποτελέσουν τον πυρήνα του προγράμματος. Είμαι ευτυχής δε που βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοι όπως και οι υποφαινόμενοι έχουν επιλέξει να ε, υπερπηδήσουν το ε, κριτήριο το γεωγραφικό. Το κύριο κριτήριο είναι η αριστεία και πρέπει να είναι η αριστεία. Το Horizon 2020 δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο συνοχής. Το έχουμε ήδη συζητήσει αυτό. Αντιθέτως, θα πρέπει να εμβαθύνουμε ώστε να υπάρξουν περισσότερες συνέργειες για τα διαρθωτικά, με τα διαρθωτικά ταμεία. Πρόκειται για έρευνα λοιπόν και ανάπτυξη όμως όλα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να καλυφθεί η απόσταση ανάμεσα στις την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 13 και των υπόλοιπων 15. Τώρα, Επίσης θα πρέπει η έρευνα να καταλήγει σε συγκεκριμένες εφαρμογές συγκεκριμένες εφαρμογές ισορροπημένες και να αναγνωρίζουμε πως η βιομηχανία παίζει ουσιαστικό ρόλο στο οικοσύστημα της ε, καινοτομίας στους διάφορους τομείς και ότι έτσι είναι για ε, τις ε, Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει και απορροφά τα δύο τρίτα των ε, χρημάτων ε, για την έρευνα. Αυτοί ξέρουν, έχουν την τεχνογνωσία θα μπορούσα να εμβαθύνω και για τα open data και το σύστημα αξιολόγηση. Ε, θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια και με τους υπόλοιπους σκιώδη εισηγητές ε, για να φτιάξουμε ένα σαφές κείμενο με υποδείξει που θα δείχνουν και συστάσεις που θα δείχνουν ακριβώς ποιε είναι οι θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ, κυρία Βίρινγκ. Ο κύριος Δελούντο από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεση, γιατί θεωρούμε πω είναι ισορροπημένο και συμφωνούμε με την εισηγήτρια στα κεντρικά σημεία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιε πτυχέ που θέλουμε να τονίσουμε και που αντικατοπτρίζονται στι τροπολογίε μα. Στο πλαίσιο τη ε, του, συμφωνία αυτή, θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα την, στην έρευνα για τι κλιματικέ αλλαγέ και τι υποδομέ. Ιδιαίτερα επειδή οι ΙΠΑ εξετάζουν σημαντικέ ε, δημοσιονομικέ περικοπέ για τα ε, αμερικανικά ε, ερευνητικά κέντρα για το περιβάλλον. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε την έρευνα και την έρευνα που διεξάγεται από τα πανεπιστήμια. Χωρίς την κατάλληλη χρηματοδότηση αυτής της ερευνητικής βάσης, το, μελλοντικό, το ε, μελλοντικό δυναμικό ε, καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μεωθεί σημαντικά. Να αναγνωρίσουμε δε ότι όλα τα κονδύλια αυτά θα ε, σημειωθούν μόνο για σχετικές έρευνες και για έρευνες βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Θέλουμε επίσης να θυμίσουμε στα κρατημέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να, να κινηθούν ε, καταλήλως ώστε να φτάσουν το 3% ε, ΕΠΤΑ για αυτό τον προπολογισμό. Να περιμένουμε δε ότι θα προέλθει από τη βιομηχανία ε, το μεγαλύτερο κομμάτι των επενδύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταλούντε. Ο κύριος Μπορέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι τροπολογίε ε, μα ε, έχουν κατατεθεί με στόχο τη βελτίωση του project ε, για το Horizon 2020, επενδύσει για την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Στην Ευρώπη αυξάνονται οι αποστάσει και οι διαφορέ ανάμεσα στι διάφορε περιοχέ και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το συγκεκριμένο στοιχείο όταν αξιολογούμε τη δυνατότητα ενό προγράμματο να επηρεάσει με στρατηγικό τρόπο το μέλλον τη υπήρου μα. Είμαστε κοντά στο 2020, αλλά πόρο απέχουμε από τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Οι τελευταίοι δε είναι χώρες ε, που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να αποκλειστούν, γιατί αυτό το σύστημα ε, δίνει την προτεραιότητα και ωφελεί περισσότερο αυτούς που ήδη έχουν εμπειρία και τεχνογνωσία. Με την τροπολογία μας 63 που θέλει να μπει στην παράγραφο 8 της έκθεσης θέλουμε να τονίσουμε αυτό το πρόβλημα και να ζητήσουμε πιο ίση κατανομή των πόρων γεωγραφικά και την εισαγωγή ενός μίνιμουμ μάλλον μέγιστου κατοφλίου χρηματοδότησης που θα μπορεί να πάρει ένα συγκεκριμένος ε, ε, δικαιούχος ε, σε ένα ή σε περισσότερα χρόνια για ένα project. Εδώ εντάσσεται και η τροπολογία 92 που ζητά ενίσχυση του δικτύου επαφών σε εθνικό επίπεδο ώστε να είναι εγγυημένο και για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις η κατάλληλη υπηρεσία στήριξης στις φάσεις προετοιμασίας υποψηφιότητας. Και έτσι κλείνω και αναφέρω ένα σημείο που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές, αυτό των μικρομεσαίων. Ε, το πρόγραμμα Horizon 2020 έχει ε, είναι μάλλον ένα συγκεκριμένο ε, εργαλείο, αλλά θα πρέπει να μπορέσει και να επηρεάσει. Θέλουμε λοιπόν να αυξηθεί η γραμμή και επειδή αυξάνονται τα project ε, τα οποία ενώ περνάνε από την επιλογή μετά δεν διαλυλοποιούνται γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Αξιολόγηση λοιπόν των προτάσεων. Θέλουμε αυτό το κριτήριο να μπορεί να είναι η δυνατότητα μιας επιχείρησης να δημιουργήσει επενδύσεις και θέσεις απασχόλησης και όχι μόνο στο να μπορέσει να φέρει επισφαλή κεφάλαια έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε ποιε είναι οι εταιρείε που μπορούν όντως να το πράξουν αυτό. Τώρα, ο ετών πρέπει να κατανοήσει ολόκληρη τη διαδικασία τη αξιολόγηση, γιατί μόνο έτσι ένα επιχειρηματία μπορεί να συνειδητοποιήσει ποια είναι τα όρια και, τα, και οι δυνατότητε τη προτασή του και να μπορέσει και να τη βελτιώσει στη συνέχεια. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Έλφ για το ίδιο θέμα. Καταρχάς, να ευχαριστώ την εισηγήτρια γιατί έκανε, μιλάκι για την αναθεώρηση του ε, ορίζοντα 2020 και απ' την άλλη πρέπει να, κάνει και την, να ορίσει τη θέση του Κοινοβουλίου για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, θέλω να μιλήσω εγώ λίγο για το μέλλον και να αναφέρω διάφορα πράγματα. Καταρχάς πρέπει να δούμε σε όλα αυτά τα θέματα που θέλουμε να καλύψουμε, ποια είναι τα χρήματα που έχουμε και ποιο είναι το μοντέλο που θέλουμε να προωθήσουμε και σε ποια σχέση υπάρχει το καλύτερο δυνατό μοντέλο. Μπορούμε ας πούμε να έχουμε πολλά θέματα, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μικρότερη συμμετοχή. Ε, και αυτό τι σημαίνει, στο τελευταίο πρόγραμμα πλαίσιο, το 7, το κόστος για μη εγκεκριμένε αιτήσει από τι διάφορες επιχειρήσεις ήταν τα μισά από τα χρήματα που είχαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, οπότε αν είμαστε κάτω από το 10% έγκρισης δηλαδή, ε, θα είναι πραγματικά παράλογο αυτό, γιατί μιλάμε για τεράστιο κόστος που ουσιαστικά θα αντικατοπτρίζει ένα πολύ μικρό ποσοστό προγραμμάτων. Ε, θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια του επόμενου πλαισίου, προγράμματος πλαισίου να το σκεφτούμε αυτό. Αν δούμε δηλαδή αν θέλουμε 125% προώθηση της μεγάλης βιομηχανίας για τέτοια project ή να επικεντρωθούμε στα συγκεκριμένα προγράμματα ή να έχουμε περισσότερα χρήματα για τα προγράμματα. Πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε. Επίσης κάτι άλλο που υπόθηκε είναι το θέμα της αριστείας ως βασικής αρχής και τις δύο προκλήσεις ε, της ισορροπίας των, της συμμετοχής των φύλων και της κατανομής μεταξύ των κρατών μελών του, των διαρρών κενών που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Συχνά λέω ότι όταν ένα project ε, εγκρίνεται και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι το καλύτερο α, project, αλλά υπάρχουν και άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή των κριτηρίων, αυτό θεωρώ ότι είναι καταστροφικό λάθο. Απ' την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να πούμε ότι δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την αριστεία και να λέμε ότι δεν θα φροντίσουμε να, έχουμε αυτό το, να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της ε, προώθησης της ε, συμμετοχής γυναικών σε τέτοια project. Έχουμε 60.000 ερευνητές ε, στην, που τους χάνουμε στην Ευρώπη και, αυτό, και η απάντησή μας είναι ότι προσπαθούν θα πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες να συνδυάσουν την, οικονομική, την επαγγελματική και την προσωπική του ζωή για να παραμείνουν στην, στο χώρο εργασίας. Οπότε, όλα όσα μπορούμε να κάνουμε, ναι να τα κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν προς όφελος ε, των, ε, της αριστείας να πούμε ότι όταν το project δεν είναι πλέον το καλύτερο, να μην το αποσύρουμε εφόσον υπάρχουν άλλα κριτήρια που μας οδηγούν σε κάτι καλύτερο. Δεν κάνουμε χάρη στους ερευνητές με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την αριστεία. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτό το κενό καινοτομία στην Ευρώπη. Πρέπει να δώσουμε παραπάνω χρήματα, πρέπει να δώσουμε παραπάνω χρήματα για την ε, έρευνα, την ε, καινοτομία, την δημιουργία καλύτερων προγραμμάτων και πρέπει να έχουμε τέτοιε πρωτοβουλίε. Το έχουμε κάνει, αλλά θα πρέπει να χρειαστούμε, θα χρειαστούμε για να γίνει αυτό καλύτερα περισσότερα χρήματα. Επίσης, η, τα ΣΔΙΤ και οι κοινέ ε, δραστηριότητε. Ε, είναι κάτι που αλλάζει το παιχνίδι αυτό και πρέπει να το προωθήσουμε. Έχουμε τα βραβεία επίση καινοτομία, τα οποία είναι πολύ ορατά, είναι πολύ, παρουσιάζονται στο κοινό με, από διάφορα θέματα και θέλουμε ναι, να έχουμε τεχνολογίε breakthrough κτλ. Οπότε χρειαζόμαστε τέτοιου είδου εργαλεία όπω τα βραβεία καινοτομία. Και επίση πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το Brexit. Θα πρέπει να το δούμε στα πλαίσια των ε, διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση να πούμε ότι θα διευρύνουμε το φάσμα και ε, τη διπλωματία της επιστήμης και εμένω σε αυτό που πάντα κάνει το Κοινοβούλιο, το fast track στην ε, καινοτομία. Έχει περάσει η εποχή που κάναμε την οργάνωση της έρευνας από πάνω προς τα κάτω. Πρέπει να, είμαστε, να είναι οριζόντια η προσέγγισή μας, να έχουμε ε, ε, ευελιξία, να έχουμε γρήγορη προσαρμογή, γιατί οι καιροί αλλάζουν γρήγορα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα καλό μέσο για τη γεωγραφική ε, ισορροπία. Δεν μπορούμε τα, μικρά κράτη-μέλη να πρέπει να περιμένουν τρία-τέσσερα ε, χρόνια όταν έχουν τρία-τέσσερα καλά προγράμματα αριστείας για να τα προωθήσουν. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτούς που μπορούν να εγγυηθούν το επίπεδο που έχουμε θέσει, το επίπεδο αριστείας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, πολύ σημαντικά όσα μας είπες, αλλά ξεπέρισες και τα πέντε λεπτά. Η κυρία Τόγια έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω την εξήμισή μου για την έργο τη κυρία Καμπεθόν Ρουίση που όπω είπαν και οι συνάδελφοι είναι εξαιρετική και θα μα ε, οδηγήσει να ε, συμβάλλουμε κι εμεί ε, με θετικό τρόπο. Όλοι γνωρίζουμε το Horizon ήταν μια από τι πιο ισχυρέ δράσει τη Ένωση, τι πιο σημαντικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και άρα έχουμε το καθήκον να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσει να λειτουργήσει και να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Ε, για την κοινωνική και την ε, οικονομική της Υπήρου μας. Πιστεύω πως είναι επίσης σημαντικό να ξεκινήσουμε από κάτι που θύμισε και η κυρία Καμπεζόν και άλλοι συνάδελφοι. Ποια είναι η εξισορρόπηση, η βέλτιστη που θέλουμε ανάμεσα στη βασική έρευνα που είναι ουσιώδης, ουσιαστική και αυτό έχει προκύψει από τα 10 χρόνια ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, το European Research Έρευνα που και βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η βασική έρευνα για τι υπόλοιπε εξελίξεις και από την άλλη πλευρά να ευνοήσουμε και την καινοτομία που είναι στοιχείο κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα χρειαστούν λοιπόν και μεγάλη πολλοί πόροι. Πρέπει λοιπόν ε, Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτήν την σχέση που δεν είναι εύκολη και δεν είναι ξεκάθαρη ανάμεσα στις επενδύσεις για την πανεπιστημιακή έρευνα και την άμεση σχέση με τις βιομηχανίες για την αξιολόγηση ακριβώς αυτής της έρευνας ε, από εμπορική άποψη. Κάτι ακόμα που πρέπει να κατανοήσουμε καλά είναι οι προτεραιότητε τη έρευνα. Γνωρίζουμε ότι έχουμε όλα διάφορα προγράμματα, όλε τι διαδικασίε ε, τη Κομισιόν με το πρόγραμμα εργασία τη από χρόνο σε χρόνο και κάθε δύο χρόνια, κάθε διετία ε, ορίζονται τα προγράμματα και θα πρέπει να ακούσει περισσότερο τη γνώμη μα στο Κοινοβουλίου, όχι μόνο με αυτό το Κοινοβούλιο και να ξέρει και ποιο είναι η προτεραιότητά μας. Το σπουδαίο θέμα τη γύρανση ε, του ευρωπαϊκού πληθυσμού, α πούμε, είναι πολύ σημαντικό θέμα και όλα τα θέματα για τη, της υγείας εν ολίγηση, τις παιδικές ε, ασθένειες, ε, ο παιδικός καρκίνος. Ε, οφείλουμε να παρέμβουμε στην έρευνα λοιπόν για την υγεία και προωθώντας π.χ. δίκτυα και πλατφόρμες επαφής για αυτά τα Ινστιτούτα τα υγειονομικά που είναι κάτι το θετικό για την Ευρώπη. Και ίσως η να πρέπει να αναλάβει να συντονίσει και να οθήσει στο συντονισμό, γιατί ακριβώς έτσι θα μπορέσει η έρευνά μας ε, να φτάνει σε μεγέθη σημαντικά και να φτάσει σε ε, σημαντικά αποτελέσματα παράλληλα όπως γίνεται αλλού. Τώρα, πιο συγκεκριμένα στοιχεία, ορισμένες στοιχείες που αφορούν τη διαδικασία που για μας όμως είναι σημαντικά. Θα τα παραθέσω γρήγορα γρήγορα. Πρώτα είπε ένα συνάδελφος και εγώ το συμφωνώ μαζί του ότι οφείλουμε και πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν και από όλους όσοι κάνουν την επιλογή πρώτον να δηλώνουν εκ των προτέρων ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης. Συχνά δεν γνωρίζουν ποια είναι τα στοιχεία τα ευαίσθητα για την αξιολόγηση. για να μπορεί ο ξελογητή επί της ουσίας, ε, ε, αλλά και ο υποψήφιος επί της ουσίας να διορθωθεί για την επόμενη φορά, για να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια και να υπάρχει και αιτιολόγηση. Ένα άλλο σημείο είναι αυτό ε, επίλυση ενό προβλήματο που δεν έχουμε ποτέ μπορέσει να λύσουμε. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ερευνητικά κέντρα τα οποία οργάνονται ε, ε, συνδέονται με διακυβερνητικέ ε, οργανώσει, α πούμε, εφαρμοσμένοι φυσικοί στη Τριέστη, στη Τεριέστη, στην Ιταλία, όπου δεν μπορούν να αποσυνδεθούν. Είναι πραγματικά διαμάντια σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποια από αυτά τα ερευνητικά κέντρα. Τέλο, το είπε ήδη κάποιο. Μόνο ένα πράγμα στοιχεία, τα δεδομένα. Όχι μόνο θα πρέπει να υπάρχει πιο ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά θα πρέπει να ευνοηθεί η επανεπεξεργασία των δεδομένων της έρευνας. Υπάρχουν ένα σωρό δεδομένα τα οποία φτάνουν μέχρι ένα σημείο για την έρευνα. Δεν πρέπει να ξαναρχίσουμε από το μηδέν. Πρέπει να μπορούμε να επανεπεξεργαστούμε τα δεδομένα που υπάρχουν. Γιατί είναι ένα ακόμα ε, σκαλά και ένα βήμα μπροστά. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί τα περισσότερα ήδη υπόθηκαν. Καλωσορίζω την έκθεση της εισηγήτριας που είναι εξαιρετικά καλή και υπογραμμίζει την μεταρρύθμιση στην οποία θέλει να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο με τον οποίο δίνει έμφαση στα όσα λέει και σαφώς οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και η πίεση στον προπολογισμό σε αυτό το τομέα κομμάτι της απόδειξης της σημασίας ε, του ορίζον 2020 και είναι και ε, ενδείξεις για το τι πρέπει να γίνει περαιτέρω για την ενίσχυση του προπολογισμού και επίσης ε, να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι έχει ενταχθεί εδώ το θέμα του φίλου. η παραπομπή στο ψήφισμα του 2015 αλλά και η αναφορά στο θέμα του γένους του φίλου. Ευχαριστώ κυρία Μούντι και εγώ έβαλα τον εαυτό μου στον κατάλογο των ομιλητών διότι θέλω να κάνω τα... κάποια γενικά σχόλια. Το πρώτο είναι ότι δεν θα λειτουργήσει αυτό η υπόθεση αν ε, τα κράτη-μέλη δεν φτάσουν τον στόχο του 3%. Η Ένωση πόρο απέχει από το στόχο του 3%. Κάποιες χώρες είναι πολύ πιο μπροστά, αλλά περισσότερες είναι πίσω. Και αυτό πρέπει να το θυμίσουμε στις ε, χώρες ε, όντως να μπορέσουν να φτάσουν αυτό το στόχο. Και μια άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι υπήρχε μια παγκόσμια, ένα παγκο, παγκόσμια πορεία για την, επιστήμη, την επιστήμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ συμμετείχα στο Βερολίνο, ήταν περίπου 12.000 κόσμος οι διαδηλωτές ε, αλλά πραγματικά λυπούμε πως υπάρχει μια τάση ε, ε, να ανοείται τα απορίσματα της επιστημονικής εργασίας. Εναλλακτικά στοιχεία είναι αυτά που αντικαθιστούν τις αποδείξεις τις επιστημονικές και πρέπει να σας πω πως δυστυχώς έχουμε, εγώ έχω πολλά προσωπικά ε, μάλλον παραδείγματα αυτού του γεγονότος εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Αν εμείς εδώ, σε αυτή την Επιτροπή δεν το καταπολεμήσουμε αυτό, τότε ποιος θα το κάνει. Και γι' αυτό θέλω να κάνω έκκληση, να καταπολεμήσουμε αυτή την τάση που υπάρχει, να παραμελεί κανείς και να αγνοεί τις επιστημονικές αποδείξεις σε ένα σωρό τομείς. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις ο κύριος Βάντεμπεργκ από την DG Έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου μας δίνετε το λόγο. Είμαστε ευγνώμονες για τη μόνιμη υποστήριξη που λαμβάνουμε από το Κοινοβούλιο. Και... Όντως το Horizon 2020 είναι επιτυχές πρόγραμμα. Βλέπουμε αυτό από το μεγάλο ανταπόκριση που έχουμε από τους ενδιαφερόμενους φορείς στην δημόσια διαβούλευση αλλά και με τα πορίσματα μας που θα δημοσιευθούν στα τέλη Μαΐου θα δείξουμε ότι το Horizon 2000 ε, ε, προχωρά στην επιτύχηση των στόχων του. Ε, θα σας δώσουμε και πολύ εκτεταμένα στοιχεία και αποδείξεις πράγμα που θα οδηγήσει στο να εμποδίσουν με ε, να επικρατήσουν εναλλακτικά στοιχεία για το Horizon 2020. Ασχολούμαστε με πολλά θέματα που αναφέρατε τη συμμετοχή της βιομηχανίας, την ετοιμότητα της τεχνολογίας, ε, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις έναντι δανείων και ένα σωρό άλλα ζητήματα που θίξατε κι εσείς. Προσβλέπω στην έκθεση της εισηγήτριας και της τροπολογίας το τελικό δηλαδή αποτέλεσμα θα το λάβουμε φυσικά υπόψη και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ε, εκτιμούμε πολύ τη συνένεση που προκύπτει ότι δηλαδή πρέπει να εστιάσουμε στην αριστεία και αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λήθος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία. Επίσης καλωσορίζουμε την έμφαση στη διαφάνεια και το άνοιγμα προς όλους τους δυνατούς φορείς, την οικονομία και την κοινωνία που μπορούν και που κάνουν καθημερινά οδηγούν στην επιτυχία του Horizon 2020. Είμαστε περήφανοι που 50% των συμμετεχόντων στο Horizon 2020 είναι νεοφερμένοι σε σχέση με το προηγούμενο δηλαδή πρόγραμμα πλαίσιο και γι' αυτό θέλουμε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης αυτής στην έρευνα και στην καινοτομία. Αντίκτυπος για τις επιστήμες αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το ε, ζωντανό σας ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Και εσείς που ακούσατε τόσα καλά λόγια, έχουμε ε, τη δυνατότητα να σας δώσουμε το λόγο για να κλείσετε. Και εγώ είναι πολύ σύντομα να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και για τις καλές σας συμβολές που ήταν όλες επικοδομητικές και ενδιαφέρουσες και κυρίως για τον τόνο με τον οποίο μιλήσατε γιατί τονίστηκε ακριβώς η σημασία αυτού του προγράμματος για το μέλλον της Ευρώπης. Ακριβώς αυτήν ε, την καλή ατμόσφαιρα θέλω να διατηρήσουμε μέχρι ότου να κλείσουμε την εργασία και να βγει μια έκθεση που θα εκπροσωπεί όλες τις ομάδες ε, και το πιο σημαντικό είναι ο Horizon 2020 να διατηρήσει αυτή τη μοναδική φύση και τη σημασία του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή ε, συνεδρίαση του πρωινού δηλαδή, θα διεξαχθεί ψηφοφορία επί του κειμένου αυτού τον Μάιο, 29 και 30, στη συνάντησή μας εκείνη, εκείνη του διημέρου. Ευχαριστώ πολύ.